L'ordre Λοιπόν, σύμφωνα... Σύμφωνα με την ε, απλουστευμένη διαδικασία θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Κώστα για την σύναψη συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση τη ασφαλή πολιτική αεροπορία. πολιτικής Ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την πρώτη έκθεση του κύριου Κώστα. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορία. Υιοθετήθηκε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα ψηφίσουμε με απλουστευμένη διαδικασία την έκθεση της κυρίας Βόλης για το κοινό καθεστώς για την εμπορία ο αλβουμίνη και γάλακτα αλβουμίνη. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη θα ψηφίσουμε σύμφωνα με απλουστευμένη διαδικασία την έκθεση κυρίας Γουόλης για το φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγέ μενοχών που αφορούν εταιρείε διαφορετικών κρατών μελών καθώς για τη φορά της κρατικής έδρας αρχίζει ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Υιοθετήθηκε και αυτή έκθεση του κυρίου Μποτόπουλου για το γλωσσικό καθεστώ που ισχύει στι αιτήσει ανέρεση κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσια Διοίκηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορία υιοθετήθηκε. Έκθεση του κυρίου Μπέλτερ για τις οικονομικές ε, και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Έκθεση της κυρίας Γκίνας, της κυρίας Μαγκίνας μάλλον, για την κοινή γεωρική πολιτική και την παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε έκθεση κυρίας Γκραμπόφσκα για τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, ονομαστική ψηφοφορία. Απ. ο κύριος Μπίσλη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ονομαστικές ψηφοφορίες που είναι λίγο περίεργο για μένα, διότι πραγματικά ε, δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω ψηφίσει ναι και ψηφίζω ναι, αλλά να έρθει και ένας μηχανικός να μου το διορθώσει το μηχάνημα, σας παρακαλώ. Θα σας στείλουμε έναν τεχνικό αμέσως. Αλλά μήπως να βρείτε και καμία καινή, ε, θέση, ε, μήπως το τυχόν και λειτουργεί το μηχάνημα εκεί. Έκθεση της κυρίας Γκραμπόφσκα και ονομαστική ψηφοφορία αρχίζουμε τώρα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας υιοθετήθηκε. Έκθεση της κυρίας Βέιλερ για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Έκθεση της κυρίας του κύριου Γκερέρο για την προσέγγιση διαχείρισης της αλίας με βάση το οικοσύστημα. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζουμε. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κλάς. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. 292 ψήφια πετούνται. Εξετάζουμε την κοινή θέση Ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο κομμάτι των τροπολογιών. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Εγκρίνεται η κοινή θέση όπως έχει τροποποιηθεί. Τώρα περνάμε σε δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης ε, του Συμβουλίου για την διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Η μία τροπολογία έχει γίνει απαράδεκτη, εξετάζουμε την κοινή θέση και εδώ απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έκθεση κυρίας Μπρέγερ. Η πρώτη ομάδα τροπολογιών. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρες ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Τώρα. Τροπολογία 46. Άρθρο 4, παράγραφος 7. Τροπολογία 46 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ε, τροπολογία 178. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε το δεύτερο κομμάτι της, ε, της τροπολογίας 198. 169, τροπολογία 169, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε το αντίστοιχο κομμάτι της τροπολογίας 178 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Τώρα περνάμε στην κοινή θέση ε, όπως έχει τροποποιηθεί, η οποία υιοθετήθηκε. Πάμε στην έκθεση ε, Cleans για το συντονισμό των νομοθετικών... Α, από ό,τι φαίνεται ήταν μεγάλη επιτυχία. Και περνάμε τώρα στην έκθεση κλίνση για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες θα εξετάζουμε την πρόταση οδηγίας, ψηφίζουμε την πρώτη ομάδα τροπολογιών. Δεν υπάρχει, δεν έχει ζητήσει κανεί ονομαστική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, ε, αποχές, υιοθετείται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία θα ε, ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία και συγχαρητήριο στους συζητητές μας. Έκθεση κυρίας Γκοτάρντι, δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ, 2007 και 2008 πρόταση ψηφίσματος. Τρει τροπολογίες τη εισηγήτρια, τις ψηφίζουμε από κοινού, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Κύριο Σίλτον Χάρη, συζητάει το λόγο. Πρόεδρε, έχω την εξή παράκληση. Έχουμε στις φαραγυρικές μας συνεδριάσεις πάντα στη μέση του, της αίθουσας μία ε, κάμερα τηλεοπτική, έναν φακό. Δεν είναι βέβαια εύκολη δουλειά των κάμεραμεν, αλλά ταυτόχρονα και για τους βουλευτές δεν είναι εύκολο να δουλεύουμε όταν έχουμε στη μέση της αίθουσας μια κάμερα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε κάπως τη διαρρύθμιση της αίθουσας ή να βρεθεί μια τεχνική λύση διαφορετική, εν πάση περιπτώσει καλύτερη. Η πρόεδρος, βεβαίως, θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Χίτον Χάρης χιστής το λόγο όμως. Κύριε Χίτον Χάρης. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Διαδικαστικό. Προσπαθώ να βρεθει μια τεχνικη λυση διαφορετικη εν παση περιπτωσει καλυτερη η προεδρος βεβαιως θα απευθυνθουμε στις αρμοδιες αρχες ο κυριος χιτον χαρης χιστης το λογο ομως κυριε χιτον χαρι ναι προεδρε ευχαριστω διαδικαστικο προσπαθω να τραβηξω την προσοχή ενό κλητήρα εδώ και ώρα κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών για να δώσω τι επεξηγήσει μου, για να εγγραφώ. Αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα δεν έχει φτάσει κανεί εδώ από του κλητήρε γιατί το ρεύμα είναι προ την άλλη μεριά, προ την αντίθετη κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν δύο επεξηγήσει ψήφου γραπτέ να δώσω για την έκθεση Μπρέγερ. Παρακαλώ. Κύριε Χίτον Χάρης. En règle générale, on s'inscrit avant εν γέννη καταγραφώ, ε, εγγραφόμαστε μάλλον για τι επεξηγήσει ψήφου πριν από την έναξη των ψηφοφοριών κύριε Χιτον Χάρη, αλλά ευχαριστώ να σημειώσουμε τι επεξηγήσει ψήφου σα θα τι δεχθούμε χωρί αντίρρηση. Κυρία Ντόιλ, το αυτό, Πρόεδρε. Και εγώ παρακαλώ για την ανοχή σας, γιατί και εγώ έχω αποστείλει ε, επεξήγηση ψήφου που δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια σας. Βεβαίως, κυρία Ντόιλ, χωρίς πρόβλημα, θα δεχθούμε και τη δική σας. Επεξήγησης ψήφου, λοιπόν, τώρα.